περισσότερη συνοχή. Και όχι διχασμοί. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τα χθεσινά πρακτικά και τα σημερινά θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο προς έγκριση στην αρχή της επόμενης συνόδου. Αν δεν έχετε διατηρήσεις θα διαβιβάσω τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν σήμερα στους ε, αρμοδίους ε, φορείς και πρόσωπα που είναι οι αποδέκτες τους. Διακόπτεται η σύνοδος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λίγη συνεδρία.